So. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, περνούμε στις ψηφοφορίες τώρα. Έκθεση Τάιν. Ε, πρόκειται για το πρωτόκολλο για τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Τάιν έχει το λόγο, η συγγήτρια. Αξιότιμοι συνάδελφοι, δύο τεχνικές εκθέσεις για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι προς ψηφοφορία και διαπαραταξιακά κάνω την εξής παρατήρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ζητεί να αναγνωριστεί η αύξηση του αριθμού των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η πρόταση αυτή ε, δεν πέρασε διότι δεν μπόρεσαν τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν ε, σχετικά με την προέλευση των ε, πρόσθετων δικαστών παρόλο που υπήρχαν πολλές προτάσεις επιτάπητος. Εδώ ε, σε τεχνικό επίπεδο είχαμε μία ιδιόμορφη περίπτωση χωρίς προηγούμενο. Θα πρέπει να απαλλάξουμε τουλάχιστον εν μέρη το δικαστήριο, να με την πρόταση κανονισμού και για το πρώτο μέρος και το άλλο μέρος βέβαια, το πιο σημαντικό, ε, μένει σε εκκρεμότητα και ελπίζω μέχρι το 2013 να ολοκληρωθεί επιτυχώς και αυτό. Εξ ονόματος των πολιτών και των επιχειρήσεων καλό τα κράτη-μέλη να μην παίζουν τα συνήθη παιχνίδια τους ε, με την τρίτη εξουσία και να επιδείξουν προς αυτήν τον προσήκοντα σεβασμό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τάιν. Η ψηφοφορία θα γίνει ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Πόσελτ, βρήκατε την κάρτα σας. Μάλιστα. Εψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Πέρας. Δεκτή. Προχωρούμε. Το επόμενο μέρος για τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Εψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Μάλιστα. Πέρας λοιπόν της ψηφοφορίας. Δεκτή. Προχωρούμε στην έκθεση του κυρίου Φέρμ «Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας». Καταρχήν, όλη η ενότητα 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτά. Δεύτερη ενότητα καταπίπτει. Ψηφίζουμε τώρα στην πρόταση της Κομισιόν όσοι τροποποιήθη υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό και σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, ονομαστική ψηφοφορία εδώ, άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Συγχαρητήρια στους εισηγητές, την κυρία Τάιν και τον κύριο Φέρμ. Προχωρούμε. Έκθεση της κυρίας Μπαλσάνη, σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 3. Ψηφίζουμε καταρχήν όλο το κείμενο 1 έως 7 unblock υπέρ, κατά, αποχές, δεκτά. Το ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία στο σύνολό του, άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Μάλιστα. Πέρας. Δεκτή λοιπόν. Προχωρούμε τώρα πολιτική της Ένωσης για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ψηφίζομαι το, η πρόταση της ομάδας ECR 69 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κοινό ψήφισμα S&D, ALDE, Πράσινη και ΓΟΕ υπέρ Α, μισό λεπτό πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά το σημείο 12 12 πρώτο μέρος του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές δεκτό το πρώτο μέρος δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές αυτό θα το ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν όλοι πέρας δεκτό και το δεύτερο τώρα ψηφίζω με το σημείο 1 Τροπολογία της ομάδας ΕΛΚ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεκτή η τροπολογία. Α, έλεγχος. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Είχε γίνει δεκτό. Περνούμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος εν συνόλο. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. δεκτή η πρόταση ψηφίσματος. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά. Αυτή είναι η τελευταία μας σύνοδος πριν από τις θερινές διακοπές. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, σε όσους πάνε διακοπές.